Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τη συζήτηση αυτή. Και προχωρούμε γρήγορα στο επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη και έχουμε καθυστερήσει κιόλα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που περίμεναν υπομονετικά για να συζητηθεί το θέμα τους. Ε, είναι το σημείο υπαριθμών 6, η πέμπτη έκθεση της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, COSI. Ξέρετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 71 της συνθήκης επευλήθη η έκθεση αυτή και το άρθρο 6.2 της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής Κόζη το Δεκέμβριο. Στόχος της έκθεσης είναι η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια επισκόπηση για τις διαδικασίες που καλύπτουν στην περίοδο Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2017. Υπάρχει και μια πρόβλεψη για τον κύκλο πολιτικής 2018-2021. Κύριε Σιτάρσκα θα μας κάνει την παρουσίαση, εκπροσωπεί τη Βουλγαρική Προεδρία. Παρευρίσκεται. Παρακαλώ. Γεια σας και καλώς ορίσατε. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο εκπροσωπείτε και τον πρόεδρο της Κόζη που δυστυχώ κολλείται και δεν παρευρίσκεται. Παρακαλώ, έχουμε καθυστερήσει και σας ζητώ συγγνώμη. Θα μπορούσατε να είστε σύντομοι και είμαι βέβαιος ότι μπορείτε. Πέντε, δέκα λεπτά, παρακαλώ την παρουσίασή σας και μετά θα έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Κατανοώ ότι έχετε ε, μεγάλο πεδίο δραστηριοτήτων και εμείς Επιτροπή ε, Είναι για μένα προνόμιο η ευκαιρία που έχω να σας ενημερώσω ε, ως πρόεδρος της ε, Υποστηρικτικής Επιτροπής ΚΟΖΗ και αντιπρόεδρος της ΚΟΖΗ γιατί τι γίνεται με αυτή την επιχειρησιακή συνεργασία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Ε, έκθεση και προτεραιότητες. Λάβατε την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι γνωρίζετε τις βασικές αναλύσεις και τα ευρήματα. Θα είμαι σύντομη σε ό,τι αφορά τη γενική παρουσίαση της έκθεσης ε, και το ίδιο της το περιεχόμενο. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την έκθεση, υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της ανανεωμένη στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια, υψηλές προτεραιότητες όπως η αντιμετώπιση τρομοκρατίας, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, διαλειτουργικότητα, νέος κύκλος πολιτικής για την καταπολέμηση διεθνούς οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, ε, συνέχιση του κύκλου 2014-2017 και προετοιμασία του νέου κύκλου 2018-2021, και βελτίωση των δεσμών ε, και των σχέσεων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Η εφαρμογή της νέας ανανεωμένης στρατηγικής ασφαλείας ε, ήταν ένα θέμα που κυριάρχησε ξανά και ξανά. Η ΚΟΖΗ σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από ε, πληροφορίες από τα κράτη-μέλη έχει ελέγξει κατά πόσο και παρακολουθεί κατά πόσο όλα αυτά υλοποιούνται ομαλά. Έχουν αρχίσει και συ ζητήσεις ε, για τη νέα περίοδο. Σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία και μέτρα αντιμετώπιση, τη, αυτά παραμένουν ε, προτεραιότητα στις διαδικασίες Επιτροπή Κόζη, εξακολουθεί να παρακολουθεί την υλοποίηση των ε, μέτρων του Συμβουλίου της 20 Νοεμβρίου 2015 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 17 και 18 12 του 2015. Οι τρομοκρατικέ επιθέσεις εντόπισαν αδυναμίες στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια, που κατά προτεραιότητα έπρεπε να διορθωθούν. α πούμε η διαχείριση της πληροφορία και διαλειτουργικότητα συστήματων πληροφοριών για την ασφάλεια των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια. Η ανταλλαγή λοιπόν των πληροφοριών και η διαχείρισή τους ήταν σημαντική και προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις 9 και 10 Ιουνίου του 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα δικό χάρτη για την ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών ε, και τα λοιπά σε τομέα εσωτερικών και δικαιοσύνης. Επίσης το αντίστοιχο Συμβούλιο 8 και 9 Μαρτίου, ενιστώ τους έχους, ε, ε, επιβεβαίωσαν και οι Υπουργοί τη σημασία που αποδίδουν στα πλαίσια των νομοθετικών προτάσεων που έχουμε επιτάπητο στο θέμα αυτό. Επίσης, η Επιτροπή Κόζεν έκρινε ε, την ε, εφαρμογή και υλοποίηση του οδικού χάρτη και έχει αναφέρει και αναθέσει ε, κάποια θέματα που πρέπει να εξετάσουν πυρογνώμονες, ομάδα εργασίας τρομογλωτίες και ΣΥΣ-ΣΥΡΕΝΕ. Χρειάζεται μια προσέγγιση στην καταπολέμηση της δημοκρατίας διαρθρωμένη και ε, πολυεπίπεδη και πολυτομεακή. Ε, ε το αντίστοιχο έγγραφο έχει συμπεριληφθεί στην έκτη ε, μηνιαία έκθεση. Στα πλαίσια αυτά η ΚΟΣ επίσης συζήτησε την ενίσχυση συνεργασίας για την καταπολέμηση της δημοκρατίας και την ανάλυση απειλής. Είναι δυνατό να μην τα διαβάζετε με τέτοια ηλικιώδη ταχύτητα για να σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Θα τα πω πιο αργά. Και ζητώ συγγνώμη για το ρυθμό, την ταχύτητά μου. Έλεγα λοιπόν, ενίσχυση συνεργασία στην καταπολέμηση της απειλής ε, της τρομοκρατίας και ανάλυση της απειλής ε, γίνονται διάφορες προτάσεις για συνολική αντιμετώπιση της εικόνας της απειλής και εκτίμηση αυτής. Ε, αυτά τα προετοιμάζουν τα αντίστοιχα παρασκευαστικά όργανα. Γίνονται εκθέσεις για την εκτίμηση απειλής τρομοκρατίας με κάποιες συστάσεις και συμπεράσματα για πολιτική στα αντίστοιχα όργανα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη τον συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στην ΚΟΣ. Σε ό,τι αφορά το νέο κύκλο τώρα πολιτικής 2016, το τρέχοντα μάλλον 2017, ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος γιατί Είχαμε πάρα πολλές δράσεις για την υλοποίηση του κύκλου 2014-2017 και την προετοιμασία του νέου κύκλου 2018 2021. Εξακολουθεί η Κόζη να παίζει ε, πρωταγωνιστικό ρόλο. εξάμεινο παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και όλου του κύκλου πολιτικής 2014-2017 και μετά από τις διάφορες εκθέσεις των εμπειρογνωμών των εθνικών συντονιστών και ε, των υπολείπων και της Ευρωπόλ κάνει συστάσεις στα πλαίσια τώρα ε, του κύκλου πολιτικής θα πρέπει να τονιστεί και κάτι ακόμα. Οι επιδόσεις των κοινών ε, ημερίδων δράσης. Τι σημαίνει αυτό. Έχει γίνει πολλή δουλειά το τελευταίο διάστημα έτσι ώστε να συνενωθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των κοινών ημερίδων δράσης στα κράτη-μέλη ε, σε συντονισμό με την Ευρωπόλ. Θέλετε να σας δώσω ένα ε, παράδειγμα επιτυχίας. Τον Ιούνιο 2017 είχαμε μια παγκόσμια ημερίδα δράσης για τους αερολιμένες. για την ε, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων με ε, κλεμμένες ή πλαστές πιστοτικές κάρτες. 153 ύποπτοι λοιπόν συνελήφθησαν, στα σύνορα, 312 συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές έχουν εντοπιστεί και άλλες συνδέσεις με άλλα εγκλήματα. Έχουμε λοιπόν ετήσιες ε, στρατηγικές ε, κατευθυντήριες γραμμές που συνδέονται με τις ημέρες δράσης, ημέρες μάλλον, για την, το σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των δράσεων αυτών από κοινού. Το 2016 η ΚΟΖΗ επίσης συμφώνησε για τον ορισμό των κοινών δράσεων στις μέρες αυτές για να βελτιωθεί η επίδοση το 2017, πράγμα που έγινε. Επίσης, πρωταγωνίστησε η Κόζη στην στρατηγική καθοδήγηση στο θέμα της χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανομή και τη χάραξη προτεραιοτήτων στους πόρους ε, που έχουν ε, αφιερωθεί στις προτεραιότητες. Ξέρετε από την έκθεση ότι γίνεται και αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα το 2017 έγινε αυτή και τα ευρήματά της χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να σχεδιαστεί ο νέος κύκλος πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2018-2021. Η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης των νέων προτεραιοτήτων άρχισε το Μάρτιο του 2017 στην Κόζη όταν η Επιτροπή έλαβε γνώση της ε, εκτίμησης απειλής σόκτα για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Ε, το παρουσίασε αυτό η Europol. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και άλλες στρατηγικά έγγραφα, εκτιμήσεις και πολιτικές και έχει καταλήξει σε 10 προτεραιότητες για τον επόμενο κύκλο. Ε, κυβερνοχώρος, ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, παράνομη μετανάστευση, οργανωμένο έγκλημα ιδιοκτησίας, ε, ε φοροδιαφυγή ε, σε δασμούς, ε, λαθρεμπόρες, πυροβόλα όπλα, παραχάραξη, πλαστογράφηση εγγράφο, περιβαλλοντικά εγκλήματα. Είναι 10 οι προτεραιότητες αυτές για το 2018-2021 και τον αντίστοιχο κύκλο πολιτική. Εγκρίθηκε το Μάιο του 2017. Και τέλο, κατά την περίοδο αυτή, η ΚΟΖΟ επίση συμφώνησε του όρου αναφορά του νέου κύκλου πολιτική. Τι σημαίνει αυτό. Εκεί υπάρχουν τα βασικά στοιχεία, βήματα και άλλα στοιχεία της πολιτικής. Κοινά σχέδια δράσης, επιχειρησιακά προγράμματα και λοιπές ε, δραστηριότητες. Αν σας ενδιαφέρει μπορώ να σας ενημερώσω ε, και ε, για άλλες εργασίες της Επιτροπής Κόζη. Κατά το τελευταίο 1,5 χρόνο αυτό ε, που μας απασχόλησε ήταν να συνδεθεί εξωτερική με την εσωτερική ασφάλεια και ενίσχυση της ασφάλειας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος ε, Να συνεχίσω ή να σταματήσω εδώ. Προτίμησα αυτά τα 15 λεπτά να σας κάνω μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση, αλλά θα συνεχίσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις αν θέλετε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Όπως μπορείτε να δείτε, πολύ λίγοι συνάδελφοι είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, ζητήσατε το λόγο. Σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η εκπρόσωπος της Βουλγαρικής Προεδρίας, πολλές φορές εμείς αναφέραμε ότι για θέματα εσωτερικής ασφαλείας έχουμε πρόβλημα και κυρίως με τη μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και εγκληματικότητα μεταξύ αυτών των ε, μεταναστών που ζητούν βοήθεια ακόμη και αυτοί οι οποίοι παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια που προσπαθούν να διασώσουν ζωές στη θάλασσα. Επίσης διώκονται. Οι Ισπανοί διώκονται σχεδόν παντού. Ακόμη και στην Ελλάδα. Διότι ενώ παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια Συγχαίρεται η... τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες, τα θέματα της ιστορικής ασφάλειας. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε κάπως αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λόπες, θέσατε το θέμα σας και εγώ θα ήθελα επίσης ενα παρεμφερές θέμα να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, στα πλαίσια της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, διότι αυτά υπογραμμίστηκαν ως προτεραιότητες στον τομέα της εγκληματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του πολιτικού κύκλου 18-21. Και βεβαίως αυτό μας μας απασχολεί όλος ιδιαίτερο στην Επιτροπή μας. Κυρία Ευχαριστώ, Κλώτ. Είναι πολύ στενή δική μου ερώτηση. Γιατί δεν κατάλαβα καλά αν η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανήκει ως θέμα στις αρμοδιότητες σε όλα αυτά που μας παρουσιάσατε. Γιατί θα ήθελα κάποια σχόλια σε σχέση με την Cambridge Analytica είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την λειτουργία, την εύρυθμη της δημοκρατίας μας και τους κινδύνους. Τι προβλέπετε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στάρσκα. Θέλετε σύντομα να δώσετε απαντήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. για το θέμα της ε, προτεραιότητας ως προς την παράδειγμα, Ο Πρόεδρος, με συγχωρείτε, είχε στήσει η κυρία Σπινέλη το λόγο. Αν μου επιτρέπετε να ακούσουμε και αυτή την ερώτηση και στο συγγνώμη σας διακόπτω. Κυρία Σπινέλη. Θέλω να προσθέσω κάνα δύο πραγματάκια κι εγώ. Για το μεταναστευτικό πάλι, την παράτυπη μετανάστευση. τους πράτους μετανάστευσης που, μετα... που αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, απατεώνες και κτλ. Και ανησυχώ ιδιαίτερος διότι ένας πρόσφυγας που ζητάει άσυλο προσπαθεί να ξεφύγει από μια εμπόλεμη ζώνη εξορισμού είναι παράτυπος μετανάστες. Άρα και σε αυτόν τον ορισμό έχουμε πρόβλημα. Δεύτερο, το ερώτημα της κυρίας Κέντζε για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και θα ήθελα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, παρακαλώ. Για τους όρους συλλογής δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα και αν ε, γίνεται σεβαστό Τόσο στο σύνολο του οικονομισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ναι, λέει ο πρόεδρος, αν θέλετε, μιλήστε πρώτα για το θέμα αυτό της μετανάστευσης και μετά για τα προσωπικά δεδομένα. Δύο είναι τα θέματα σας. Ναι, ευχαριστώ. επιχειρησιακό σχέδιο παράτυπη μετανάστευση. Ως πεδίο, ως αντικείμενο έχει κυρίως τα δίκτυα των λαθροδιακινητών μεταναστών. Αυτό για να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση στην, ε, αυτού του είδους του εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε τα τελευταία χρόνια σημαντικά εγκλήματα και φρονομώ ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας στο πεδίο αυτό έχουμε να κάνουμε δηλαδή με εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν μετανάστες παραβιάζοντας τα δικαιώματα και βέβαια τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Τα τελευταία χρόνια η COSI και η GHA έχουν επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα και δίνουν αποφασιστικές απαντήσεις στην ε, πρόκληση αυτή περιθώριο για παρερμηνίες ή παρεξηγήσεις εδώ δεν βλέπω, γιατί η διακίνηση μεταναστών είναι έγκλημα, μπορεί να έχει, να έχει και σημαντικό κίνδυνο και πάντως παραβιάζει τα δικαιώματα των ε, μεταναστών. Ως προς την σύμπτωση ε, μεταξύ της λαθροδιακίνησης και της παράτυπης μετανάστευσης, καταρχάς έχουμε μια πολυτομιακή προσέγγιση και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Europol και οι υπηρεσίε που διαχειρίζονται τα τρία διαφορετικά κεφάλαια έχουν μια συντονισμένη συνεργασία και κοινέ δράσεις όπου βλέπουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως ε, ίσως να γίνεται διακίνηση ανθρώπων σε συνδυασμό με παράτυπη μετανάστευση. Ο πρόεδρο πριν περάσετε στο θέμα για το In Cambridge Analytica, θέλω να επισημάνω ότι όλη αυτή η σύγχυση έχει να κάνει και γιατί και καταλαβαίνουμε ότι είναι προτεραιότητα η διακίνηση ανθρώπων, αλλά ε, όλη αυτή η σύγχυση οφείλεται στο γεγονό ότι αυτό, αυτή η κλιματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ω παράτυπη μετανάστευση. Επομένως, ε, εκεί πέρα υπάρχει ο λόγος ε, της σύγχυσης. Το είπαν και οι δύο συνάδελφοι και παρακαλώ να επισημανθεί από πλευρά τη ΛΥΒΕ πω ε, η παράτυπη μετανάστευση δεν, είναι, δεν συνιστά έγκλημα αυτή αυτή. Μπορώ να είμαι έτσι ομό και απερίφραστο και παρακαλώ να ξανακοιτάξετε την ορολογία που χρησιμοποιείτε. Γιατί χαρακτηρίζεται ω προτεραιότητα καταπολέμηση εγκλημάτων ε, στο εγγύ μέλλον. Θέλετε να περάσετε στο θέμα της Cambridge Analytica. Ναι, ευχαριστώ. Για διευκρίνηση όμως από πλευράς μου. Ο όρος ολόκληρος είναι καταπολέμηση της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης. Επομένως εδώ έχουμε να κάνουμε με, τους, με τα δίκτυα των διακινητών. Εκείνων που καταχρώνται, που παίρνουν χρήματα από το μετανάστη που του προσφέρουν μέσα ταξιδίου επικίνδυνα. Και προσπαθούμε να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση και να καταπολεμούμε αυτό το φαινόμενο που έχει να κάνει με τη διακίνηση και την εκμετάλλευση του μετανάστη. Προστασία δεδομένων. Εδώ δεν είναι συγκεκριμένο κομμάτι της δουλειάς της ε, ΚΟΖΗ. Έχουμε να κάνουμε ένα εγκάρσιο θέμα που εφαρμόζεται σε κάθε τομέα της δουλειάς μας. Η συλλογή δεδομένων, πληροφοριών. Για κάθε κανόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως η οδηγία για τις αστυνομικές αρχές έχει δώσει ιδιαίτερη θέση στο θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα συμπεράσματα για το πώς μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όχι μόνο γίνεται σεβαστή, αλλά ε, τη χάνει και ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμού και επιτήρηση προς την εφαρμογή της από την κόζη για την υπόθεση Cambridge Analytica. Την εξετάζουμε όχι τόσο συνέπειες για την κόζη, όσο για τη δουλειά των διαφορών υπηρεσιών της. Γιατί η κόζη έχει αναλάβει επιχειρησιακά το στρατηγικό συντονισμό, δηλαδή πρόκειται για συγκεκριμένε επιχειρησιακές προσεγγίσεις και όχι για συγκεκριμένε υποθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη δουλειά τη κόζη. Αν σα ενδιαφέρει πάντω, έχουμε να κάνουμε με ένα πλαίσιο πολιτικής που καθοδηγεί τι εθνικέ αρχές. Στο πλαίσιο της κόζη το παρακολουθούμε και λαμβάνουμε υπόψη την εφαρμογή του όταν έχει σχέση με τις δραστηριότητε μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, ότι κάποια στιγμή θα συζητήσουμε το θέμα αυτό της Cambridge Analytica και όλα τα στοιχεία μας προσθέτω. Ευχαριστώ κυρία Σιτάρφη, καθώς και την ομάδα σας μέρους της Προεδρίας της Βουλγαρίας. Συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στο οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι το 1745 το θέμα της αποστολής στην Σλοβακία. 6Q2, and that's at 17.45. Jan 6Q2, and that's the, um, the draft delegation report on Slovakia, um, which I know some colleagues are interested in. So 6Q2 at 17.45. Λοιπόν, 17 και 45 θα ε, συνεχίσουμε τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην αίθουσα 6Q2.